θα λάβουν το λόγο οι συντάκτες των ψηφισμάτων για το θέμα αυτό. Ο κύριος Σεμπαστιά είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας ε, για τη συνένεση, το συμβασμό ε, για το κοινό αυτό ψήφισμα. Είναι ένα μακροσκελές πολύπλοκο ψήφισμα, κάτι πολύπλοκο, μάλλον αναπόφευκτο όταν μιλάμε για την Αιθιοπία. Αυτό που θέλουμε να καταγγείλουμε εδώ είναι η καταστολή εκ μέρους της κυβέρνησης κατά ειρηνικών διαδηλωτών, αγροτών, οι οποίοι καταδικάζουν τις προσπάθειες επέκτασης ε, του Μητροπολιτικού Κέντρου της Αντίς Αμπέμπα διότι έτσι ε, θα επιδεινωθούν ε, οι φυσικές καταστροφές. Είδαμε πώς υπέρμαχοι ανθρωπίνων δικαιωμάτων να διώκονται με 140 τουλάχιστον νεκρούς. Είναι κατεπήγον το θέμα και γι' αυτό το συζητούμε σε αυτό το πλαίσιο αλλά θέλαμε να πλαισιώσουμε το ψήφισμα αυτό, γι' αυτό είναι και τόσο μακροσκελές, αναφέροντας τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αιθιοπία. Μια χώρα με αποτυχημένη ε, δημοκρατία, ε, που είναι όμοιρος ε, ενός κόμματος που είναι στην εξουσία, που ασκεί καταστολή στους Ρώμου, στους Ογκαρέν και σε άλλες εθνοτικές μειονότητες καταστολή. Πολλοί φεύγουν και οι δημοσιογράφοι. Έχουμε αντιτρομοκρατικό νόμο, φήμος της ελευθερίας, αυθαίρετες ε, προσαγωγές ε, και δίωξη μέλων ε, των ΜΚΟ και μέχρι και πολίτες της Ένωσης είναι κρατούμενοι στις αιθιοπικές φυλακές. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαιτήσει να δοθεί δέουσα προσοχή και να τηρηθούν όλα τα διατάγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Αιθιοπία είναι και μια από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο. Όσοι έχουμε πάει εκεί έχουμε δει τέτοια επίπεδα εξαθλίωσης που δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να, να ξεπεραστούν. Η Ένωση είναι ο πρώτος χορηγός, ο πρώτος χρηματοδότης και θα πρέπει ε, να ε, εκμεταλλευτούμε ε, αυτό το ρόλο για να ε, επηρεάσουμε την κατάσταση στην Αιθιοπία. Αλλιώς δεν θα είμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Αντινόλφη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ελευθερία εκφραστή είναι θεμελιώδες δικαίωμα και πρέπει να προστατεύεται όπως προβλέπει και ε, η Συμφωνία της Κοτονού και η Χάρτα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε δεν υπάρχει κομματική δημοκρατία. Θα πρέπει αμέσως να ξεκινήσει πολιτικός διάλογος με συμμετοχή όλων, ένας διάλογος διαφάνεια μεταξύ όλων των πολιτικών εκπροσώπων, με εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών και του πολίτε. Η Αφρικανική Ήπειρος είναι υπέροχη με ανεξάρτητους πόρους. Όμως πληρώνει ακόμη το τίμημα της αγριότητας της αποικιοκρατίας. Θα πρέπει εδώ λοιπόν οι Ευρωπαίοι να υποστηρίξουν του Αφρικανούς στην προσπάθεια να χειρεφετηθούν και να απαλλαχθούν από τα εμπορικά συμφέροντα και την υποβιέτηση χωρί νέε μορφέ αποικιοκρατίας και ε, την υποδήλωσή του ε, στην οικονομία των ελεύθερων συναλλαγών. Ευχαριστούμε κύριε Αντινόβλφη. Ο κύριος Ντεμεσμέκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι εθνοτικές ομάδες όπως η Ρώμο και η Αμχάρα είναι θύματα εθνοτικής βίας στη χώρα. Παρόλο τα πηγαίνει καλά ως προς την οικονομική ανάπτυξη και την ανθρώπινη ανάπτυξη, τις κοινωνικές δηλαδή προτεραιότητες η χώρα αυτή, είναι από τους καλύτερους μαθητές της Αφρικανικής Ε, είναι πρόβλημα οι εθνοτικές εντάσεις και αυτό είναι το μειονέκτημα της ε, δράσης της κυβέρνησης. Η ανεξάρτητη δημοσιογραφία δεν μπορεί να ασκηθεί στην ε, ε, Αιθιοπία ελεύθερα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τον αντίκτυπο που έχουν όλα αυτά στον πληθυσμό όπως το πρόγραμμα η πρωτεύουσα Αντίς Αμπέμπα να επεκταθεί στα δημοτικά της όρια στην περιοχή της Ομχαρίας. Αυτό έχει οδηγήσει και θα οδηγήσει ενδεχομένως την έξωση γεωργών και ένα μεγάλο μέρος του τοπικού πληθυσμού. Η κατάστασή τους είναι επισφαλής, επισφαλής παρόλο τα προγράμματα αυτά ακυρώθηκαν και επέστρεψαν στις αιστείες τους. Θα πρέπει λοιπόν να επιτελεστεί συγκεκριμένη πρόοδος και να αλλάξει η μορφή του διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε η κυρία Μπεσέρα Μπαστερετσέα. Με συγχωρείτε. Ο κύριος Πόσπισιλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόμα της ομάδας μας θα ήθελα να υποστηρίξω αυτό το ψήφισμα. Συζητάμε ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αιθιοπία και πάλι μετά από κάποιους μήνες γιατί λαμβάνω χώρα κάποια πράγματα στην Αιθιοπία. Πέρσι είχαμε πάνω από 140 άτομα τα οποία εσφάγισαν βιαίως όταν διαδηλώνανε ειρηνικά στην Αντισαμπέμπα. Τα άτομα αυτά, ε, μέλη ενός ε, μιας εθνοτικής ομάδας, αγωνιζόντουσαν κατά της αλλαγής του χωροταξικού σχεδίου της ε, Αντίσα που θα οδηγούσε σε εκδίωξή τους από τα σπίτια τους. Η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αιθιοπία χειροτερεύει και γι' αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε και πάλι αυτή τη χώρα ως ε, ενδιαφερόμενη για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ φανερό ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί στεναρά κατά τη συμπεριφορά της Αιθιοπική κυβέρνηση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει την αντιπολίτευση, της φυλάξης των ηγετών, της αντιπολίτευσης, της αντιμετώπισης των ελευθέρων μέσων ενημέρωσης, την καταστολή της ελευθερίας έκφρασης, γιατί η Αιτιοπία είναι μία από τις δέκα χώρες όπου υπάρχει μεγαλύτερη καταπίεση των, δημο, των ε, δημοσιογράφων. Υπάρχουν ακτιβιστές που πετάγονται στη φυλακή κάθε τόσο. Είναι τέτοια η νομοθεσία λοιπόν που δεν μπορεί κανείς να, δεν μπορεί κανείς να συμμετέχει σε μη κυβερνητικές οργανώσεις ή σε μη ε, κερδοσκοπικές ε, διαδικασίες. Χρειαζόμαστε, χρειάζεται η Αιθιοπία λοιπόν τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτή η βοήθεια θα πρέπει να συνδέεται με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη χώρα αυτή, να τους βοηθήσουμε, αλλά μόνο αν η κυβέρνησή τους βελτιώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ε, τώρα η κυρία Στέρα Μπαστρετσέα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μεταξύ των κρατών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια αδυναμία να κατανείμουν 160.000 πρόσφυγες μέσα σε 500 εκατομμύρια. Ενώ η Αιθιοπία αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 70.000 πρόσφυγες από την Ερυθρέα, από το Σουδάν και άλλες περιοχές και είναι συγχρόνως και πηγή μεταναστών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν μονάχα με κοινή δράση για τη, για τη ρίζα του προβλήματος μετανάστες. Εγώ χαίρομαι για τη συμφωνία που επιτέφθη τον προηγούμενο Δεκέμβριο για ένα κοινό ταμείο για την Αφρική που θα δώσει 253 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδε ενέργειες, ιδίω για το κέρδο τη Αφρική, Κάτι το οποίο με απασχολεί κύριε Μιμίτσα. Ποιο είναι ο ρόλο του Κοινοβουλίου στο πρόγραμμα αυτό. Και επίσης στο ψήφισμά μας τονίζουμε ότι η Αιθιοπία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεταξύ 2014 και 2020 το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, ε, ε θα δώσει 748 εκατομμύρια. <clears throat> Υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε τα κονδύλια αυτά να μην καταλήξουν να υποστηρίζουν την ε, καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Η κυρία Βελζιά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και 10 χρόνια αυτό είναι το πρώτο ψήφισμα για την Αιθιοπία και γι' αυτό είναι και τόσο μακροσκελές. Από το 2009 όμως υπάρχει τμήμα καταστολής ε, φήμος των ελευθεριών, αυθαίρετες ε, προσαγωγές, ε, ποινικοποίηση ΛΟΑΔ, εξοδικαστικές εκτελέσεις πολλοί ε, αγρότες ε, επειδή μπορεί να τους ε, διώξουν από τις γέες τους έχουν ξεσηκωθεί. Επίσης, μεγαλύτερη εδώ και 50 χρόνια ξηρασία βιώνει η χώρα και διαγράφεται ο εφιάλτης μιας ανθρωπιστικής καταστροφής. 5 εκατομμύρια παιδιά είναι σε κατάσταση απόλυτης ανάγκης. Σίγουρα υπάρχουν μεταναστευτικές πιέσεις από τις γειτονικές χώρες και όλες οι χώρες περιοχής ε, αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Με τη διαδικασία του Χαρτούμ ε, υπάρχουν ε, οι προϋποθέσεις για μια νέα πολιτική, όμως αμφιβάλλω για το πώς θα χειριστεί η Ευρώπη αυτά τα κύματα των προσφύγων κάθε ε, εταιρική σχέση θα πρέπει να έχει ρήτρε για βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προσφύγων. Πρέπει να υπάρξει πρόσωπο μεγαλύτερη δημοκρατία. Είναι κατεπήγον το θέμα τη Αιθιοπία. Έχει η Ένωση προωθήσει το σεβασμό της ε, πολιτιστικής ε, ποικιλομορφία της Αιθιοπία, που είναι και μια, ένας από του μεγαλύτερου από του μεγαλύτερους της Ευχαριστώ. Κύριος Αντώνιο, Πιέρα Αντώνιο Παντσέρη, τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Εδώ και κάποιους μήνες στην Αιθιοπία και στην Ορομία υπάρχουν ε, προβλήματα με τα όρια της δημοτικής με τα δημοτικά όρια της πρωτεύουσα της Αντίς Αμπέμπα. Το έχουμε εντοπίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη είχαν προκληθεί προβλήματα στους ντόπιου γεωργούς, διότι δεν μπορούσαν να ασκήσουν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους και ζούσαν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. 140 διαμαρτυρώμενοι ε, διαδηλωτές ε, δολοφονήθηκαν και πάρα πολλοί άλλοι ε, φυλακίστηκαν από τι δυνάμει ασφαλεία. Από το 2005 επισημαίνουμε την επισφαλή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Όλε αυτέ οι μορφέ εχθροπραξία, μορφέ βία πρέπει να πάυσουν, καθώ και παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικέ φυλακίσει. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε την αφοσίωση τη Αιθιοπία στην ε, συνεργασία τη με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα προσφύγων και μεταναστών, αλλά θα πρέπει να ξαναδούμε και την παρακολούθηση τη βία από την αιθιοπική κυβέρνηση και το κατά πόσο υπάρχουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της χώρας όπως ε, το πλήθυσμα μας ε, εντοπίζει. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Παντζέρη και τώρα εκπροσώπη των πολιτικών ομάδων πρώτη από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες η κυρία Γκόμες. Η καταστολή των διαδηλωτών στην Αντίς Αμπέμπα οδήγησε σε 140 θανάτους και είναι η πιο πρόσφατη απόδειξη της πολιτικής ομότητας και βίας οποιαδήποτε ε, ζωντανή αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης. Υπάρχει καταστολή και παρακολούθηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ε, αυτό ισχύει για τους ειρηνικούς διαδηλωτές και τους ε, ειρηνικούς αντιφρονούντες. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ανάπτυξη απαιτούν να μην παραποιούνται στατιστικά δεδομένα που προβλέπουν την αρπαγή γεών ώστε να αυξηθούν τα δημοτικά όρια της πρωτεύουσα χωρίς να ε, λαμβάνονται υπόψη ανάγκες των ανθρώπων στην Ρωμία και αλλού στη χώρα. Θα πρέπει λοιπόν οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση με όλα τα κράτη-μέλη να μην στηρίζουν τον προπολογισμό για να συνεχίζει την καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η νόμιμη κυβέρνηση. Πρέπει να δούμε τη σταθερότητα ολόκληρη αυτή τη γεωγραφική περιοχή. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι οι αρχέ και οι αξίε ε, δεν γίνονται σεβαστές και αυτό ε, οξύνει την αστάθεια και τις αντιπαραθέσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ολόκληρη αποσταθεροποίηση την Αφρικανική Ήπειρο. Ξέρουμε τι έγινε με την Αραβική Άνοιξε από το 2011. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρχει σεβασμός της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αιθιοπία. Έφτασε επιτέλους αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριο Γιακόφ Τσίτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. είναι μακρός ο κατάλογος των αντιδημοκρατικών ενεργειών της ε, Αιθιοπία. Λυπούμαστε γιατί είναι μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου συγχρόνως, όμως αυτός ο κατάλογος, ο οποίο <clears throat> περιλαμβάνει και κατάχρηση της αντιτρομοκρατική ομοθεσίας για να καταπιέζει την ε, αντιπολίτευση, τους δημοσιογράφους και γενικά όλους τους πολίτες της χώρας και όλες τις μειονότητες στην ε, Αιθιοπία δεν είναι κάτι που μπορούμε να αποδεχτούμε. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το χωροταξικό σχέδιο ανάπτυξης της, της Αμπέμπα αντιστοιχεί σε αρπαγή γης από την περιοχή των Ρωμαία. Γι' αυτό ζητούμε από την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να ξεκινήσει ένα διάλογο μαζί μας και με τον ΟΗΕ για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να δίνουμε βοήθεια στην Αιθιοπία που είναι μια χώρα που χρειάζεται βοήθεια. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, η κυρία Παλώμα Λοπέ Βερμπέχο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τις ομάδες που, <clears throat> τις πολιτικές ομάδες της κοινή του για να καταδικάσουμε την ε, καταστολή στην ε, Αιθιοπία και για να καταγγείλουμε την οικονομική και πολιτική κατάσταση στο κέντρο της Αφρικής που έχουν οδηγήσει σε ένα ρεύμα από πάνω από 700.000 πρόσφυγες στην περιοχή. Πρέπει να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή, αυτή την κατάσταση, να ελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι και να εξασφαλιστεί ο πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά η ευρωπαϊκή ευθύνη ξεπερνάει μονάχα αυτέ τι εκκλήσει. Πρέπει, που είναι κατεπίγουσε, υπάρχουν οικονομικέ ευθύνε. Η συμπερίληψη τη Αιθιοπίας στο παγκόσμιο εμπόριο και οι πολυεθνικές εδρεώνουν την ανισότητα και την έλλειψη πρόσβασης στη γη. Καταδικάζουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στην ένδια και στην έλλειψη κοινωνικών δικαιωμάτων. Πρέπει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να μην χρησιμοποιούν τρίτες χώρες ως φυλακές, ενώ συγχρόνως απεμπολούν τις ευθύνες τους για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανησυχούμε γιατί αναπτυξιακά κονδύλια χρησιμοποιούνται για την εσωτερική καταστολή και όχι για την ανάπτυξη σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Θα πρέπει εκεί να δώσουμε την προτεραιότητα και όχι μονάχα να είναι μονάχα μια συνοδευτική ενέργεια όπως θέλει να το κάνει η Κομισιόν. Ευχαριστούμε. Ο κύριος τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Αιθιοπία εκπροσωπή έναν από τους πιο αρχαίους ε, πλούσιους ε, πολιτισμούς ε. και υπάρχουν άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών που συμβίωσαν επί αιώνες. Όμως τα τελευταία χρόνια επιδεινώνεται σοβαρή κατάσταση, πολλαπλές παραβιάσεις των δικαιωμάτων, κοινωνικο-οικονομική πρόοδος στη χώρα έχει ανασταλεί τα πρόσφατα γεγονότα στην ε, ε, χώρα με τις προσπάθειες επέκτασης της Αντισαμπέμπα οδήγησαν σε ακόμη περισσότερες παραβιάσεις, ε, παρενόχληση της αντιπολίτευσης, ε, φήμωση των μέσων ε, μαζικής ενημέρωσης και καταστολή των ΜΚΟ. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ε, μείζον ε, χρηματοδότης, παρέχει βοήθεια στην Αιθιοπία και θα πρέπει να αναβαθμίσει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της κατάστασης με κάθε ε, μέσο που έχει στη διάθεσή της. Η Αιθιοπία μπορεί, έχει τις δυνατότητες να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που είναι σήμερα. Και εμεί πρέπει να δίνουμε χείρα βοηθεία. Η κατάσταση αυτή δεν είναι ευεργετική προ κανέναν και θα πρέπει να αλλάξει το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ. Διαδικασία Catch the Eye. Κύριος Πόλτσακ, ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι πεπισμένος ότι η καταστολή απέναντι σε αντιφρονούντες πολιτικούς κρατουμένους, δημοσιογράφους, η κατάσταση φτώχεια δεν δίνει μια καλή εικόνα για τη χώρα και σίγουρα ε, είναι τεράστιος και ο αντίκτυπος. Ίσως και η προσφυγική κρίση να είναι απλά ε, η κορυφή του παγόβουνου. Όμως πρέπει ξεκάθαρα να υπενθυμίσουμε στις αρχές Αιθιοπίας ότι η κυβέρνηση ε, θα πρέπει να είναι η κυβέρνηση μιας δημοκρατικής χώρας έχει παρέλθει η εποχή των αυτοκρατοριών. Και πρέπει να τα καταγγείλουμε όλα αυτά και να δείξουμε και τι μπορούμε να κάνουμε και μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας. Χωσέ Γνάθιο Φαρία. Ο επόμενος. Τους τελευταίους δέκα μήνες έχει σκοτώσει η κυβέρνηση Αιθιοπίας 140 άτομα που διαδηλώναν η ειρηνικά στην πρωτεύουσα Αντισαμπέμπα κατά της αρπαγής των αγροτικών γεών τους για το χωροταξικό σχέδιο της Αντισαμπέμπα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που ακολουθεί τον φόνο 56 φοιτητών που είχαν διαδηλώσει πριν από 5 χρόνια το 2011 για το θέμα αυτό. Και η κυρία Μογκερίνη έχει ήδη ζητήσει να υπάρξει μια λύση ειρηνική για αυτήν την σύγκρουση. Την ε, προηγούμενη εβδομάδα <coughs> το κυβέρνηση της Αιθιοπίας είπε ότι θα αποσύρει αυτό το σχέδιο συμβολή για την επίτευξη κάποιες συνδιαλέγειες. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε όμως ότι αυτό το τέχνασμα θα μας γελάσει. Εμείς θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αρθώσουμε το ανάστημά μας κατά της πολιτικής αυτής της αιθιοπικής κυβέρνησης. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Επίτροπος ε, Μίμητσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κάτι μέλη της έχουν έναν συστηματικό και ειλικρινή διάλογο με την κυβέρνηση της Αιθιοπίας για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, υπάρχει ένα μήνυμα που παραλαμβάνεται ότι η οικονομική και η κοινωνική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζουν με τι ε, πολιτικέ ελευθερίε και τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να είναι βιώσιμη. Μια ε, κοινωνία των πολιτών ισχυρά οργανωμένη το δικαίωμα του συνασπίζεστε, που ασκείται ελεύθερα, όλα αυτά συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί μια οικονομικά ανεξάρτητη και σταθερή χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά την ε, ε, ανησυχία και τις μορφές βίας στην Ορομία με όσα συνέβησαν γύρω από την πρωτεύουσα, την Αντίς Αμπέμπα και με μεγάλη ε, ανησυχία. Επίσης, στην Ομχαρία υπάρχει αναταραχή η οποία οδήγησε και αυτή σε απώλεια ανθρώπινων ζώων. Στις 23 Δεκεμβρίου πέρσι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει εγκρίνει ε, μία δήλωση για την ε, επίλυση της διαφοράς. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει διάλογος για να επιληθούν όλες οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν παράπονα. Οι μορφές βίας και παραβίασης που έχουν διαπραχθεί κατά των διαδηλωτών είναι περιπτώσεις για τις οποίες θα πρέπει να υπάρξει λογοδοσία. Έχουμε γύρει τις ανησυχίε μας αυτές ε, στις αιθιοπικές αρχές, προσφάτως μάλιστα στις Βρυξέλλες, όταν ο Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, όταν ο Δ. Τέντρος, ήρθε για να συναντήσει την ύπατη εκπρόσωπο, την κυρία Μογκερίνη, στις 13 Ιανουαρίου. Αναγνώρισε ότι η κατάσταση έχει έτσι και παραδέχτηκε ότι έπρεπε να ανακληθεί και να ακυρωθεί το πρόγραμμα επέκτασης των δημοτικών ορίων της Αντίσα Μπέμπα. Όμως συνεργαζόμαστε και για άλλα παρόμοια θέματα με την κυβέρνηση. Ο πληθυσμός της χώρας έχει αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες. Τώρα ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ε, αυτό είναι θέμα ε, από την άποψη της απασχόλησης, της ε, επάρκειας πόρων και της καταπολέμησης της ένδυας. Δύο συνεχόμενες περίοδοι ξηρασίας και φυσικές καταστροφές έχουν αφήσει 10,2 εκατομμύρια ανθρώπους σε κατάσταση ένδυας και ανάγκης ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπάρχουν κυβερνητικά προγράμματα που δεν εξαρκούν και αυτό εμποδίζει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει και θα συνεχίσει να παράσχει πολιτική και οικονομική συνδρομή για να προστατεύσει το, πώς, το επίπεδο προστασίας την, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αιθιοπία ταυτόχρονα και με την καταπολέμηση της ένδυας και με άλλα ανθρωπιστικά ζητήματα. Είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος του 11ου Αναπτυξιακού Προγράμματος με ένα χαρτοφυλάκιο 445 εκατομμυρίων ευρώ η Αιθιοπία όπου συμπληρώνονται με περιφερειακά και θεματικά προγράμματα και καταπιστευματικές δραστηριότητε για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων τη λάθρομετανάστευση και του εκτοπισμού πληθυσμών στην Αφρική. Παρά αυτές τις τεράστιες ανάγκες, η Αιθιοπία έχει μια πολιτική ανοιχτών θυρών και είναι η μεγαλύτερη χώρα υποδοχής προσφύγων στην Αφρική με 700.000 πρόσφυγες το λιγότερο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό θα έπρεπε να μεταφράζεται σε υποστήριξη μέσω των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης και περιφερειακής ανάπτυξης του κέρατος της Αφρικής και με το, τη συμφωνία που υπογράφηκε για την κινητικότητα και τι νόμιμε οδού μετανάστευση. Η Αιθιοπία είναι ένα σημαντικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλού τομεί. Μετανάστευση, κλιματικέ αλλαγέ, περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Για να αναφέρω μόνο μερικέ. Καλωσορίζουμε την θετική συμμετοχή της αιθιοπικής κυβέρνησης προ την Ευρώπη και αυτό βεβαίω ωφελεί και την ευρύτερη περιοχή. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με πυγμή θα συνεχίσει να τονίζει τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού του στην Αιθιοπία και να προ... παρακινεί τη χώρα να σέβεται τι θεμελιωδεί ελευθερίε όλων των πολιτών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Έχω 7 σχέδια ψηφίσματος για αυτό το θέμα. Θα κλείσουμε τώρα τη συζήτηση και η ψηφοφορία θα έπρεπε να λάβει χώρα μετά από την επόμενη συζήτηση. Σε μερικά λεπτά δηλαδή. Τελευταίο σημείο, η Βόρεια Κορέα. Ξεκινώ με τους εισηγητές παραβιάζεται εντελώς τους κανόνες. Από τους 751 έχουμε καμιά 45 αριά βουλευτές. Για διαφωτίστε μας σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς που μπαίνουμε στον κόπο να παραμείνουμε εδώ. Γιατί δεν μας δίνετε το λόγο στο πλαίσιο της διαδικασίας ΚΑΣΤΙΑΗ. Και αν αποφασίσετε, και δεν ποτέ να μην μας δώσετε τελικά το λόγο από απλή ε, συναδελφικότητα. Δεν θα έπρεπε να μας πείτε γιατί